Είμαστε αλληλέγγυοι με τους πολίτες της τσεχικής δημοκρατίας που όπως οι άλλοι ε, υπήκοοι των ε, κρατών των άλλων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα έπρεπε να μπορούν να μπαίνουν στον Καναδά χωρίς ε, βίζα. Μετά, δήλωση 2. Στις 11 Μαρτίου για 7η φορά θα γιορτάσουμε την Ευρωπαϊκή ημέρα των θυμάτων της τρομοκρατίας. Αυτή την ημέρα, το 2004, έγιναν οι βομβιστικές επιθέσεις στη Μαδρίτη και σκότωσαν περίπου 200 ανθρώπους. Και αργότερα μετά από 6 μήνες στο Λονδίνο σκοτώθηκαν 52 άνθρωποι. Δεν δικαιολογείται που δεν είναι τρομοκρατία. Καμία τρομοκρατική επίθεση, κανένας τρομοκράτης δεν θα μπορέσουν να αποδυναμώσουν το πνεύμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και της ε, δημοκρατίας. Και τώρα τρίτη πληροφορία. Έχουμε λάβει κάποιες πληροφορίες που δημιουργούν ανησυχίες όσον αφορά την επαναφορά της θανατικής ποινή στην Ταϊβάν για πέντε άτομα που περιμένουν εκτέλεση. Η επαναφορά λοιπόν της θανατικής ποινή το 2010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 να σας πω τη η διάσκεψη των Προέδρων την 5η στις 3 Μαρτίου του 2011 ενέκρινε το σχέδιο των συνόδων του προγράμματος